σε όλους. Να σας όλους τους αγκρίτους συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΠΕ. Ας επανέλθουμε στις εργασίες της τακτικής συνεδρίας Επιτροπής ΛΥΠΕ, χαιρετίζοντας τον Υπουργό, κύριο Άλαν Σάτερ, τον Ιρλανδό Υπουργό Δικαιοσύνης Ισότητας και Άμυνας και ασκούντα την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις την περισμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο καλωσορίσαμε τον Ελληνό Πρωθυπουργό, τον κύριο Γέννη, και είμαι πεπισμένος δεν θέλω να ρισκάρω υπερβολικά, αν πω ότι με μετά την παρουσία που κάνει ο κύριο Σάτερ θα τον καλωσορίσουμε και αυτό θερμά. Τον ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την καλή του διάθεση να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας για το επικείμενα εξάμεινο. Ε, κρίσιμη σημασία σε αυτή την περίοδο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι περνάμε στην τελευταία πλέον περίοδο τη θητεία μα στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε αυτό το έτο είναι καθοριστική σημασία για να ολοκληρωθούν πολλέ εργασίε ή τουλάχιστον να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά στο μέτρο του δυνατού ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πλέον σημαντικά ε, ζητήματα που εκκρεμούν. Είμαστε λοιπόν τώρα στα χέρια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Θα δώσουμε το λόγο στον Ιρλανδό Υπουργό να πάρει το λόγο να μας παρουσιάσει α, τις προτεραιότητες για ένα περίπου 15 λεπτό και μετά ως είδηστε θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων από τον Υπουργό και έπειτα μπορούν να πάρουν το λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για επιμέρους θέματα. Οπότε θα έχουμε και δεύτερο γύρο για συζήτηση. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Σάτερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα δικαιοσύνη ιστορικών υποθέσεων στην Επιτροπή σας. Παρότι είναι η 7η κατά σειρά Προεδρία της Ιρλανδίας και συμπίπτει και με την 40η επέτειο της προσχώρησής μας στην τότε ΕΟΚ, αυτή είναι η πρώτη Ιρλανδική Προεδρία όπου η δικαιοσύνη και τα εσωτερικά ζητήματα εντάσσονται στις κανονικές δομές συνθήκες και θα ε, μπορούν να συνοδευτούν από ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου. Οι κοινέ μα ευθύνε ε, είναι ευρεία κλίμακα, αγκαλιάζουν μια σειρά ζητημάτων θεμελιώδου σημασία για πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτε που ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήματα ουσιώδη για την ασφάλεια, την προστασία τους, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Όλα αυτά είναι στην καρδιά της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω στην ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συμφέρον των πολιτών μας, ώστε να προωθήσουμε την νομοθετική ατζέντα που έχουμε ενώπιόν μας. Επίσης, αυτή είναι η πρώτη φορά για την Ιρλανδική Προεδρία που θα ενταχθεί στη διαδικασία της ομάδας των τριών προεδριών. Θα προωθήσουμε την ατζέντα που πρόσφατα δημοσιεύθηκε από το πρόγραμμα της ομάδας των τριών, όπως συμφωνήθηκε από τους εταίρους μας στη Λιθουανία και Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο βασικό στόχο ε, τη 30 αυτή ή για το επόμενο 18 μήνα είναι να ενισχύσουμε το δυναμικό της Ένωση να ανταποκριθεί στις κείμενε προκλήσεις οικονομικού, χρηματοοικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η Ιρλανδική Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή όπου έχουμε μια σειρά από καταληκτικές ε, ημερομηνίες στον ορίζοντα. Το πρόγραμμα των τριών προεδριών προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος αυτού του νομοθετικού κύκλου. Και μάλιστα η πενταετής περίοδο που συμπεριλαμβάνεται από το πρόγραμμα στο Χόλμης θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2014. Βεβαίως, την παρούσα στιγμή η μεγαλύτερη ανησυχία για τους πιο πολλούς Ευρωπαίους είναι η ανάγκη για οικονομική σταθερότητα και επιστροφή στην ανάπτυξη. Δεν θα εκπλαγείτε όταν θα δείτε ότι το κεντρικό θέμα της Προεδρίας Ελληνικής εστιάζει στην σταθερότητα, θέση εργασίας και ανάπτυξη. Η πρόκληση του να επιστρέψει η οικονομία της Ευρώπης σε μια ισχυρή και σταθερή θέση που να δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασία είναι κάτι που θα κυριαρχήσει στις προσπάθειές μας κατά της προεδρίας μας. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναγνωρίσουμε και να θέσουμε τις προτεραιότητες. Εμείς, στον τομέα δικαιοσύνη ιστορικών υποθέσεων, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για να προωθήσουμε την οικονομική δραστηριότητα, την ανάπτυξη και να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία θέσεων εργασία σε όλη την Ένωση. Η ατζέντα για την δικαιοσύνη για ανάπτυξη επισημαίνει μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν για την προώθηση τη οικονομική δραστηριότητα και τη ανάπτυξη και μεταξύ αυτών ετάζονται οι κύριε προτεραιότητε τη Ιρλανδία. Προτάσει όπω ε, τα μέτρα για την προστασία δεδομένων δεν εξυπηρετούν μόνο την προστασία τη οπτική σφαίρα των Ευρωπαίων πολιτών, που είναι κάτι πολύ χρήσιμο από μόνο του, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη ε, των καταναλωτών στις ε, ε, επιγραμμικές ε, συναλλαγές και ενθαρρύνει περισσότερη χρήση τους. Αυτά τα μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του δυσνορικού εμπορίου στην ιστορική αγορά και υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, καινοτομία και εν τέλει απασχόληση σε αυτό το διοπρινόμενο χώρο. Περισσότεροι άνθρωποι που θα επιχειρούν ε, μέσω του διαδικτύου είναι καλό για την ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ψηφιακή αυτή εποχή, τα δεδομένα είναι θεμελιώδου σημασία για τόσε πολλέ καθημερινέ μα δραστηριότητε. Ο όγκος των δεδομένων στα οποία έχουμε πρόσβαση δημιουργούν μεγάλες ε, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόκληση για τις νομιστικές αρχές, ώστε να προστατεύονται τα άτομα από την κακή χρήση αυτών των δεδομένων. Παρομοίω, στην εφαρμογή του νόμου, η πρόσβαση στα ορθά δεδομένα είναι ουσιώδη σημασία για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε περίπλοκε εγκληματικέ οργανώσει, αλλά είναι και δεδομένα που ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και να διχάνουν ρυθμίσεων. Η επίτευξη προόδου στο πακέτο των δεδομένων είναι προτεραιότητα κλειδί για την ελληνική Προεδρία. Η νομοθεσία που είναι σχεδιασμένη για να μειώσει του κινδύνου για τι επιχειρήσει και ιδίω τι μικρέ επιχειρήσει που συμμετέχουν στο διασυνορικό εμπόριο έχει μεγάλο δυναμικό ώστε να αυξηθεί η δραστηριότητα και άρα να οδηγήσει σε πιο πολλές εργασίες. Τέτοια μέτρα συμπεριλαμβάνουν και την πρόταση για μια εντολή διατήρηση λογαριασμών και την πρόσφατα δημοσιευθήσα πρόταση για την αφαιρεγκαιότητα. Αυτά τα μέτρα είναι προτεραιότητα στην Προεδρία μα. και η πρόταση για έναν κοινό ευρωπαϊκό νόμο πωλήσεων ελπίζουμε να προωθηθεί. Τώρα θέλω να περάσω σε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία πιστεύω είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για την Επιτροπή σας. Πρώτα απ' όλα για την προσέγγιση δεδομένων. Ήδη ανέφερα εκδοθυγώ στην προσέγγιση δεδομένων στο πλαίσιο του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσουμε την ιδιωτική σφαίρα των Ευρωπαίων πολιτών, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ε, συναλλαγές στο διαδίκτυο και να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη χρήση και να συμβάλλει στην αύξηση του κοινωνικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά. Τώρα που θέλω να αναφερθώ στα σχέδια μας για να προωθήσουμε αυτό το μέτρο περαιτέρω. Η Προεδρία θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή για να προωθήσει το πακέτο μεταρρυθμίσεων. Προτεραιότητα που δίνουμε στην προσοχή δεδομένων ε, διαφαίνεται και το γεγονό ότι τα ζητήματα προ τα συζητήσαμε και στο άτυπο συμβούλιο Τζάι που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε μια επικοδομητική συζήτηση για μια σειρά σημαντικών θεμάτων του προτινόμενου κανονισμού, το πεδίο εφαρμογή ε, τη λεγόμενη εξαίρεση των οικοκυριών, το δικαίωμα του να ξεχαστεί κανεί και το καθεστώ διοικητικών κυρώσεων. Η προσδεδομένων δεδομένων επίσης θα είναι στην ατζέντα ε, των Συμβουλίων ε, Υπουργών ε, Τζάι το Μάρτιο και τον Ιούνιο. Η Προεδρία χαιρετίζει το, την έκθεση μάλλον στις προηγούμενες εκθέσεις που εξέδωσαν ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ε, αρμόδιες ηγητές το περασμένο μήνα και ελπίσουμε να προωθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας το κομμάτι που μας αναλογεί. Μια άλλη προτεραιότητα κλειδί για την Προεδρία είναι η οδηγία για την δέσμευση και την δίνευση των προϊόντων εγκλήματος. Στο άτυπο Συμβούλιο της προσμένης εβδομάδας οι Υπουργοί άκουσαν μια παρουσίαση από τον επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου Προσωπικών Στοιχείων Προϊόντων εγκλήματο. Σε εθνικό επίπεδο είχαμε μια επιτυχή εμπειρία στην στόχευση τέτοιων προϊόντων εγκλήματο. Τέτοια καθεστώτα δίμευση στα αστικά ζητήματα αυξάνουν όλο και πιο σημαντικά και αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του όλου τοπίου α, της ε, δήμευσης προσωπικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν ε, με τις προτάσεις μηδέας αναγνώρισης που περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχουμε αντίστοιχη πρόοδο στον τομέα των εντολών δήμευσης Και δεν θα περιοριστούμε μόνο ε, σε θέματα διήμευσης μετά από ποινικέ καταδίκες. Το Συμβούλιο κατέληξε μια γενική προσέγγιση για το σχέδιο οδηγία 7 Δεκεμβρίου 2012 και τώρα θα ξεκινήσει η διαπραγματεύση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Από ό,τι γνωρίζω, η ψήφο προσανατολισμού τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το σχέδιο οδηγία έχει αναβληθεί γιατί περιμένετε τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, ελπίζουμε σύντομα η Επιτροπή σα να είναι σε θέση να προβεί σε τη ψήφο προσανατολισμού επί τη πρόταση, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το Κοινοβούλιο να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια για να βρούμε ένα κοινό τόπο για τόσο σημαντική αυτή πρόταση. Η οδηγία για το φάκελο των ατομικών στοιχείων των ε, επιβατών αεροπλάνων είναι σημαντική δέσμευση για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το σοβαρό έγκλημα και προτεραιότητα τη Ένωση. Γι' αυτό το λόγο θα επιδιώξουμε όση πρόοδο είναι δυνατή κατά την Προεδρία μα, ώστε να υπάρξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Δεν έχω αυταπάτε. Ξέρω πόσο επίμαχαν ορισμένα θέματα στην προτινόμενη οδηγία. Τη διαφορετικότητα των απόψεων επίση γνωρίζω από διάφορε πλευρέ και τη γενική δυσχέρεια που δημιουργεί η πρόταση για το PNR για το Κοινοβούλιο και τώρα και στο παρελθόν. Ξέρω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι σε όλες τις ενασχολήσει με το θέμα αυτό θα πρέπει προτεραιότητα να είναι η ασφάλεια των πολιτών και ότι τα κράτη-μέλη τη Ένωση πρέπει να συνεργαστούν προ αυτή την κατεύθυνση. Το PNR είναι ένα μέσο που έχει αποδείξει την αξία του στην αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας για να καταπολεμήσουν τις μάστιγες ε, του λαθροπυρού ναρκωτικών, της οματεμπορίας και φυσικά της τρομοκρατίας. Όλα αυτά αποτελούν κοινέ απειλές για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, έχω επίσης πλήρη συνείδηση των ανησυχιών για την ιδιωτική σφαίρα, τον έλεγχο της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα από την αστυνομία και τις αρχές ασφαλείας και τις ανησυχίες για το εύρο τη πρόταση. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά για να καταλήξουμε στη σωστή ισορροπία για την πρόταση PNR για τους φακέλους προσωπικών δεδομένων επιβατών. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με το Σέγγεν που θα μας απασχολήσουν. Όπως ξέρετε, το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, SIS-2 όπως είναι γνωστόν, είναι ζωτική σημασία. Περιμένουμε εδώ και καιρό αυτή τη δεύτερη γενιά 2 που θα βελτιώσει το υπάρχον σύστημα, θα επιτρέψει την σύνδεση ε, συναγερμών και τον συνδυασμό βιομετρικών δεδομένων με τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Έτσι θα ενισχύσουμε την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Η επιτυχής μετάβαση από το ΣΥΣ1 στο ΣΥΣ2 κατά την Ιρλανδική Προεδρία αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κρατημέλη και την Επιτροπή για το θέμα αυτό. Η Προεδρία αισιοδοξεί ότι θα έχουμε καλά νέα να αναφέρουμε στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό τους προσεχείς μήνες. Είμαστε επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητοι για το πόσο σημαντική είναι μια ρωμαλαία και συνεκτική διακυβέρνηση του Σέγγεν, ούτω ώστε να προστατεύσουμε το κεκτημένο του Σέγγεν στο πλαίσιο αυτό. Το πακέτο για διακυβέρνηση είναι σημαντικό και για μας και για εσά. Ήδη ουσιώδη πρόοδο επετεύχθη κατά την Κυπριακή Προεδρία, ούτω ώστε να υπάρξει διακανονισμό για τα θέματα αυτά, ούτω ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανησυχίε και των δύο θεσμών. Ελπίζω το ίδιο πνεύμα συνεργασία να συνεχιστεί και να εμπνεύσει τι συζητήσει που θα γίνουν κατά τη διάρκεια τη δική μα Προεδρία, ούτω ώστε να καταλήξουμε επιτυχώ. Επίση, το θέμα τη ε, συμμετοχή τη Βουλγαρία και τη ε, Ρουμανία στο Σέγγεν ελπίζουμε να προωθηθεί κατά την Προεδρία μα. Προ το σκοπό αυτό, θα θέσω το θέμα αυτό στη μερίσια διάταξη του Τζάι τον Μάρτιο. Θέλω τώρα να σα ενημερώσω για τα σχέδια της Προεδρίας σε σχέση με την μετανάστευση, τις προξενικέ θεωρήσει και τα θέματα ασύλου. Η Προεδρία καλωσορίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κοινού συστήματος προξενικών θεωρήσεων για να τονώσουμε την ανάπτυξη. Αυτή η ανακοίνωση συνάδει πολύ καλά με τι βασικέ προτεραιότητε τη Προεδρία, ούτω ώστε να βρούμε τρόπο να έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Θα συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή για να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία με συγκεκριμένο τρόπο. Γενικό στόχο τη Προεδρία σε σχέση με τα θέματα προξενικών θεωρήσεων είναι να καταλήξουμε επιτυχώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα προξενικών θεωρήσεων όσο γίνεται και να προωθήσουμε ουσιοδός νέα θέματα. Υπάρχουν δύο άλλα θέματα που είναι ανοιχτά, που ε, διαπραγματευόμεθα με το Κοινοβούλιο και που θα ολοκληρώσουν τη δημιουργία του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου, όπω το προβλέπει το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Συγκεκριμένα, η οδηγία για τι διαδικασίε ασύλου και ο κανονισμό Ευρωντάκ. Η Προεδρία αναγνωρίζει την σημασία ολοκλήρωση στα θέματα αυτά για το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Και προ αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε μαζί σα για να επιλύσουμε τα ανοιχτά θέματα. Στόχο τη Προεδρία θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και για του δύο τομεί αυτού, ούτω ώστε να ολοκληρωθεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Σε σχέση με τον προτινόμενο κανονισμό Eurodac, είναι σημαντικό εξ αρχή να σημειώσουμε ότι το σύστημα αυτό είναι θαυμάσιο παράδειγμα συγκεκριμένη συνεργασία που να στηρίζει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου όσον αφορά την επιβολή του νόμου, δηλαδή την, καλύτερα την πρόσβαση των υπηρεσιών επιβολή του νόμου στο ΕυρωΝΤΑΚ, σημειώνουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν επί τη αρχής ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια πρόσβαση για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και άλλων σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Το Προεδρείο θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο για να επιληθούν όλα τα επίμαχα θέματα σε σχέση με τον κανονισμό αυτό, ούτω ώστε να υπάρξει επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και να είναι ακρογωνία λήθο του συστήματο ευρωπαϊκού ασύλου το κύριο θέμα που είναι ανοιχτό για τις ε, διαδικασίες του ασύλου και την οδηγία αυτή αφορά την ε, αντιμετώπιση των ετούντων άσυλων που έχουν ανάγκη ειδικών εγγυήσεων διαδικαστικών και των ε, ανηλίκων που δεν συνοδεύονται. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έχει προσφέρει ένα κείμενο για να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό, το οποίο τώρα το συζητά το Συμβούλιο. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο ανησυχεί, διότι το Συμβούλιο δεν έχει οθετήσει στην πρώτη ανάγνωση θέση για τις ε, προϋποθέσεις ε, υποδοχής και τον κανονισμό του Δουβλίνου, για τις οποίες έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ξέρω ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει υιοθέτηση, γιατί σημαντικός αριθμός κρατών μελών θα προτιμούσε αυτή τη φάση να υιοθετηθούν όλα τα ανοιχτά ακόμη θέματα μαζί. Αυτή η προτίμηση ε, μερικά προκύπτει λόγω ε, της διασύνδεσης των διαφόρων θεμάτων αυτών. Στόχος της Προεδρίας είναι να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο για να υπάρξει συμφωνία για τα εναπομένοντα στοιχεία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Πιστεύω ότι όλα τα στοιχεία του προτινούμενου συστήματος μπορούν επισήμω να υιοθετηθούν στο αρκετά εγγυσμένο. Τα μέτρα για την νόμιμη μετανάστευση θα προσπαθήσει γι' αυτά η Προεδρία να καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο για την οδηγία για του εποχιακά εργαζόμενου και του ε, μετατιθέμενου εντό των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε ότι περαιτέρω προτάσει για του ε, φοιτητέ και του ερευνητέ που θα δημοσιευθούν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα και ανάλογα με την ημερομηνία δημοσίευση θα αρχίσουμε διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για τι προτάσει αυτέ. Σε σχέση με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, MFF, μετά την καλή προπαρασκευαστική εργασία από την Κύπρο και τη Δανία, οι προτάσεις ε, τον ε, περασμένο Νοέμβρη του Προέδρου Φαν μείωσαν τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών και καταλαβαίνω ότι τώρα προχωράει δουλειά ε, και ότι ο κύριος Φαν κάνει άτυπες διαβουλεύσεις πριν επανέλθει στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τελική συμφωνία ως πρόεδρος και εθνικά η Ιρλανδία θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επαρκεί πόρου για να μπορέσει να επιτελέσει τα καθήκοντά τη σε έναν προπολογισμό που να μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση. Φυσικά, ω Προεδρία, Θέλουμε να υπάρξει ώστε να το πιο σύντομα συμφωνία. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ο πρόεδρο Φανρόμπο να έχει την επαρκή ευληγησία για το πώ θα προχωρήσει η εργασία για το θέμα αυτό. Σε σχέση με τα μέσα τζάι του πολιτού πλαισίου, η Προεδρία θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο στο μέγιστο δυνατό για να υπάρξει συμφωνία. Κατά την Προεδρία μα, η Ιρλανδία θα δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που υποστηρίζουν το δικαίωμα των πολιτών και το κράτο δικαίου. Τα δικαιώματα των πολιτών. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η οδηγία για το δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο στι ποινικέ δίκες. Στόχο Προεδρίας είναι να υπάρξει συμφωνία με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Δεν κάλυψε όλα τα θέματα που ε, περιμένει η Προεδρία να την απασχολήσουν στα πλαίσια του Τζάι. Ελπίζω όμω να χορήγησα στην Επιτροπή σα μια σφαιρική επισκόπηση των προτεραιοτήτων μα στον τομέα Τζάι σε σχέση με τι αρμοδιότητες τη Επιτροπή σα. Για άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, ε, είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα που είχα να κάνω αυτή την παρουσίαση και ελπίζω να την βρήκατε ενημερωτική. Όπως είπα από την αρχή, προσβλέπω στη συνεργασία σας και στη συνεργασία συνολικά με το Κοινοβούλιο και βεβαίω με χαρά να απαντήσω στις ιεσδήποτε ερωτήσεις σας με όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Σάτερ για την παρουσίαση. Και τώρα Αρχίζει ο πρώτος γύρος συζητήσεων με τους συντονιστές εξ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και μετά θα υπάρξει δεύτερος γύρος για τους υπόλοιπους βουλευτάς. Ο συντονιστής του ΕΛΚ, Γιώργος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισήγησή σας και την παρουσίασή σας. Δεν ήμουν βέβαιος αν θα μιλούσατε και για την ε, μετανάστευση γιατί είστε υπουργό δικαιοσύνη, αλλά ευτυχώς το κάνατε. Η Προεδρία σας έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και βέβαια στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε με θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για, τους θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά τους επόμενους μήνες και αναμένουμε πολλά από την Προεδρία σας. Χαίρομαι γιατί που είπατε ότι θα ασχοληθείτε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται με το θέμα του Σέγγεν. Γνωρίζουμε και εσείς και εμείς τα θέματα, τα προβλήματα εκεί, ότι πέντε εκθέσεις έχουν παγώσει στο Κοινοβούλιο, διότι η διαθεσμική λειτουργία της Ένωσης δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε οι αποφάσεις του Συμβουλίου δηλαδή πριν από μερικούς μήνες απέτρεψαν τη διεκπαιρέωση των εκθέσεων. Το Κοινοβούλιο μας επιμένει ότι πρέπει να βρεθεί κάποιο συμβιβασμός, κάποια εξισορρόπηση, κάποιος τρόπος να σεβαστούμε επιτέλους τη συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως τις ρήτρε που αφορούν το θέμα αυτό για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και για το μέλλον. Από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι βλέπουμε από την Προεδρία σας, Αρχικά θετική είναι η προσέγγιση μας, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε κάτι παραπάνω ως προς το πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Βέβαια αναμένουμε επίσης από την Προεδρία σας να καταλήξει και η δέσμη για το άσυλο που για μας είναι πολύ ενδιαφέρον και προκλητικό θέμα. Πιστεύουμε ότι καιρός είναι η Ευρώπη να έχει κοινέ διατάξεις ολόκληρη